δικαιωμάτων της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και το πρώτο θέμα είναι η θρησκευτική ελευθερία στο Πακιστάν. Συντάκτες Πρώτος ο κύριος Τάνοκ για ένα λεπτό. Um, η αδυναμία του Πακιστάν να αναπτύξει μια ισχυρή δημοκρατία έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ε, ανεξιθρησκεία στη χώρα αυτή για να δικαιολογήσουν την ε, καταπίεση των ε, μειονοτήτων και την ε, αυταρχικότητα ιδιαίτερα του στρατού έχουν κάνει πολλές προσπάθειες. Το Σύνταγμα του Πακιστάν στηρίζει την θρησκεία αλλά αντίθετα ισχύουν οι θρησκευτικοί νόμοι που, είναι, που επιφέρουν διακρίσεις κατά των μη μουσουλμάνων και των μειονοτήτων. Το θέμα της ε, θρησκευτικής ταυτότητας που ήταν ε, η βάση για το, δημιουργία του Πακιστάν δυστυχώς φαίνεται να προωθεί ένα κλίμα μη ανοχής. Η, ε, η εξάπλωση μηνυμάτων κατά της δύση έχει οδηγήσει σε ακρότητες, σε εξτρεμισμούς και πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν υποστεί τέτοιου είδους διαδηλώσεις. Η Ταλιμπάν του Πακιστάν είναι μια τρομοκρατική ε, ομάδα η οποία ε, τελευταίος ε, ε, προέβησε μια τρομοκρατική επίθεση στην Times Square των, της Νέας Υόρκης. Εμείς πιστεύουμε στην ελευθερία, στην ανεξιθρησκεία και την ισότητα. Και τώρα η κυρία Γιατερμάκη, η άλλη συγκέντρια, για ένα λεπτό επίσης. my group, welcomes Η ομάδα μας καλωσορίζει τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση του Πακιστάν από τον Νοέμβριο του 2008 υπέρ των θρησκευτικών μειονοτήτων και υποστηρίζει και τις προσπάθειες που κάνει ο αρμόδιος υπουργός ε, για τις μειονότητες για να υπάρχει ε, αρμονική συμβίωση μεταξύ των διαφόρων ε, κοινοτήτων, θρησκειών και δογμάτων και να προωθηθεί ο διάλογος. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά στο δρόμο προς μια πραγματική γνήσια θρησκευτική ελευθερία στο Πακιστάν. Μελέτες και εκθέσεις που έχουν κάνει ανεξάρτητοι φορείς δείχνουν ότι οι μειονότητες στο Πακιστάν στερούνται βασικών ε, αστικών ελευθεριών και ίσων ευκαιριών ε, στην απασχόληση, στην εκπαίδευση και την πολιτική εκπροσώπηση. Γι' αυτό οι νομικές διατάξεις είναι πάρα πολύ ε, ασαφείς, επικίνδυνα ασαφείς και παραμένουν ακρεμή ζητήματα που αφορούν πιστούς όλων των θρησκειών στο Πακιστάν. Επίσης γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες στο Πακιστάν αντιμετωπίζουν βία στην οικογένεια και σωματική και ε, ψυχολογική βία. Πρέπει να γίνουν λοιπόν πάρα πολλά. Ευχαριστώ. Η κυρία Κόρχολα, επόμενη, για ένα λεπτό επίσης. puhenainen. Pakistania koskeva päätöslauselmamme Ευχαριστώ. Ε, το ψήφισμα του Πακιστάν για τις ε, θρησκευτικές ελευθερίες είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή ε, και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον ορισμό της βλασφημίας. Η σημερινή κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει τακτική, να αλλάξει δρόμο και θέλουμε να την εθαρρύνουμε να συνεχίσει το μέλλον να τηρεί και να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Υπουργός Αβασπάτη την περασμένη εβδομάδα Συναντήθηκε και με το κόμμα μας, με το Λαϊκό Κόμμα και τον υποστηρίζουμε στις προσπάθειες μεταρρυθμίσεων που κάνει. 5% είναι η ποσόστοση για τις μειονότητες ε, στις δημόσιες θέσεις. Υπάρχει και αργία ε, ειδική που αφιερώνεται στην ελευθερία των θρησκειών. Όλα αυτά είναι καλέ προσπάθειε και θα πρέπει να τα υποστηρίξουμε, αλλά δεν θα πρέπει στου μετρεσέδε, στα θρησκευτικά σχολεία να στρατολογούνται τρομοκράτε. Ε, η πολιτική αυτή είναι η καλύτερη ε, μέθοδο να καταπολεμήσουμε και τα αίτια τη τρομοκρατία και την ίδια τη τρομοκρατία. και αν γίνει πραγματικότητα θα είναι μεγάλη υπόθεση. Η κυρία Γκέριγκερ Ντεόντεμπερκ, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είναι θέμα ελευθερίας ανεξιθρησκείας. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε πλέον αυτές τη, αυτή την άνηση μεταχείριση. Αλλιώς θα πάει το πράγμα πολύ μακριά οι διώξει και η καταπίεση των θρησκευτικών μειονοτήτων στο Πακιστάν πρέπει να καταδικαστούν. Εκτός αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 260 του Συντάγματος του Πακιστάν, οι πολίτες χωρίζονται μεταξύ μουσουλμάνων και μη μουσουλμάνων σε δύο κατηγορίες. Αυτό το λέει το Σύνταγμα και τα διαβατήρια το γράφουν. Και η κοινότητα των Αχμέντι ε, ε, καταπιέζεται και διώκεται ιδιαίτερα δεν έχει το δικαίωμα ούτε του συνέρχεσθε, ούτε να δημοσιεύει βιβλία και κείμενα. Και τους καταδικάζουν, τους διώκουν συχνά με την κατηγορία της βλασφημίας. Αυτά είναι όλα πολύ σοβαρά προβλήματα και χάρη στη συμφωνία που υπεγράφει πριν από έξι χρόνια μεταξύ Ένωσης και Πακιστάν, η χώρα αυτή θα πάρει 200 εκατομμύρια βοήθεια Πρόσφατα όμως φάνηκε ότι το Πακιστάν είναι έτοιμο για σοβαρές αλλαγές και θα ελπίζουμε σύντομα να πραγματοποιηθούν και να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μια αλλαγή προς ισότερη μεταχείριση. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κινίλσεν για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, η ανεξιθρησκεία δεν είναι κάτι που υπάρχει στο Πακιστάν. Έχουμε διαπιστώσει επανειλημμένως διώξεις και καταπίεση θρησκευτικών μειονοτήτων και πάνω από 80% του πληθυσμού των μειονοτήτων ζει στα όρια της ανέχειας. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί το μόνο πρόβλημα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Πακιστάν. Υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί στην ελευθερία του συνέρχεσθε, απειλές κατά οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συνδικαλι... η καταπίεση συνδικαλιστών και δημοσιογράφων. Από τότε που το Πακιστάν δέχτηκε την έννοια του πολέμου κατά της τρομοκρατίας, εκατοντάδες χιλιάδες ίσω άνθρωποι κατηγορούνται για σύνδεση, με τρομοκρατικέ οργανώσεις και γίνονται συλλήψει χωρί ένταλμα, κρατήσει σε κρυφά και μυστικά μέρη στη Λαχώρη, στη φυλακή της Λαχώρης διαπιστώθηκε ότι ενώ υπήρχε δυνατότητα κράτησης 1.500 εκρατούν το πάνω από 4.000, 4.691 μάλιστα. Ορισμένες γυναίκες τις καίνε. Εδώ θα χρειαζόταν δύο ώρες ολόκληρες για να σας διηγηθώ τι υφίστανται οι γυναίκες στο Πακιστάν και γι' αυτό το κοινοβούλιο μας επειδή σέβεται τα δικαιώματα των γυναικών, την ελευθερία της συνείδησης θέλει να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα που έχει της αρνησικυρίας για να μην επεκταθεί, παραταθεί η συμφωνία με το Πακιστάν εάν δεν γίνουν σεβαστοί οι όροι με τους οποίους είχαμε κατά πρώτο λόγο δεχτεί να Υπογραφή η συμφωνία αυτή. Ευχαριστούμε. Τελευταίος συντάκτης ο κύριος Higgins. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ω ε, Διεθνή Σοσιαλιστή, υπερασπίζομαι το δικαίωμα κάθε ατόμου στην ε, ε, αναξιθρησκεία και στην άσκηση τη θρησκευτική του πίστη, επί τη βάση ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των υπολείπων δεν παραβιάζονται. Ο λαό του Πακιστάν και ακόμη περισσότερο οι θρησκευτικέ μειονότητε του Πακιστάν αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένε ανάμεσα στην θρησκοληψία του πακιστανικού κράτου και Ε, στις, ε, από την άλλη πλευρά από τις ε, σκοταδιστικές δυνάμεις των Ταλιμπάν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να υποστηρίξει τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει τον πόλεμο στο Αφγανιστάν που έχει πολύ σοβαρές, σοβαρό αντίκτυπο στο Πακιστάν με πολύ επιζήμιες συνέπειες. Η σφαγή αμάχων στο Αφγανιστάν από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και από δυνάμεις και από εξοπλισμούς δυτικούς στο Πακιστάν γιατί ξέρουμε ότι πολλές από τις αντιδραστικές ομάδες χρησιμοποιούν δυτικά όπλα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν επίπεδα φτώχειας απίστευτα. Και η κυβέρνηση καθώς και το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έχουν να δώσουν απάντηση στον κόσμο. Η προοδευτική οργάνωση εργαζομένων είναι ένα, μια οργάνωση που προσπαθεί να φτιάξει, ε, να ενώσει ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες ε, σε ένα σε μια οργάνωση. Αυτό είναι, αυτό το μέλλον που θα πρέπει να ακολουθήσει το Πακιστάν. Ευχαριστώ τώρα εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων ο κύριος Πόσελτ, καταρχήν από το ΕΛΚ. Κυρία Πρόεδρε, το Πακιστάν είναι σημαντικός σύμμαχος ε, θα πρέπει να είμαστε ε, επικριτικοί αλλά και νυφάλοι. Έχει ένα ισλαμικό χαρακτήρα η χώρα, θα πρέπει να το σεβαστούμε. Ε, συστάθηκε η χώρα από τους μουσουλμάνους της Βρετανικής Ινδίας ε, ακριβώς επειδή ήταν μουσουλμάνοι. Και οι Ινδουιστές πάλι των Αγγλικών Ινδιών έφτιαξαν την Ινδία. Περί αυτού πρόκειται λοιπόν, ε, έχουν μεγάλη ανοχή στις ε, μειονότητες, ε, θα πρέπει να το υποστηρίζουμε, όχι μόνο για τους χριστιανούς, θα πρέπει να το τονίσουμε. Και για τους χριστιανούς ε, ε, θα πρέπει να είναι η Ευρώπη ε, εκεί. Είναι μια ήπειρος που αποτελείται σχεδόν 100% από χριστιανούς. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να σεβόμαστε τον ηγετικό ρόλο του Πακιστάν στον Ισλαμικό κόσμο. Συχνά ήταν πάρα πολύ επικοδομητικός ο ρόλος αυτός και μπορεί να συνεχιστεί και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Από τους φιλελευθέρους, Σάκε, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως διάφοροι συνάδελφοι τόνισαν, συχνά γίνεται κατάχρηση της νομοθεσίας ε, της θρησκευτική από τους εξτρεμιστές ώστε να βλάψουν τις μειονότητες. Φυσικά η ελευθερία της θρησκείας είναι σημαντική αλλά και η ελευθερία από τις διάφορες θρησκείες είναι σημαντική. Η, ελευθερία έκφρασης καταπιέζεται, κατα... παραβιάζεται στο όνομα της θρησκείας. Το Πακιστάν ε, απαγόρευσε ένα κοινωνικό δίκτυο εντός του Facebook. Ε, επίσης και επέβαλε σε όλους τους προμηθευτές ίντερνετ να μπλοκάρουν αυτό το, τον, τόπο. Ε, επίσης έχει γίνει, έχει γίνει πρωτοβουλία για να μην ε, χρησιμοποιούνται εικόνες του προφήτη. Απαγορεύτηκε και η δημοφιλή σειρά South Park που έκανε τέτοιες ε, παρουσιάσεις. Η... Η νέα γενιά του Πακιστάν ε, ε, έχει διαφωτιστεί μέσω του ίντερνετ. Πολλές φορές, ωστόσο, ε, το σχολικό υλικό φαίνεται να περιλαμβάνει πολλές διακρίσεις και διακριτικές συμπεριφορές θα έπρεπε όλοι να μπορούν να πούν τη γνώμη τους, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προσβάλλουν κάποιους άλλους. Οι προκλήσεις στην ελευθερία έκφρασης δεν ε, αντιμετωπίζονται μόνο στην Πακιστάν και στην Ευρώπη αντιμετωπίζουμε σοβαρές, ε, ε, σοβαρά προβλήματα. Ε, όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης ε, η αυτολογοκρισία γίνεται όλο και πιο σοβαρή οι ε, απειλές δέχονται οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι που εκφράζουν την άποψή τους Σας υποστηρίξουμε την ελευθερία έκφρασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Πακιστάν αλλά και σε ολόκληρο το κόσμο το καλύτερο φάρμακο κατά του εξτρεμισμού Ο κύριος Πορέμπα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι, οι εκλογές του 2008 επανέφεραν τη δημοκρατία η οποία όμως δεν είναι πλήρης στο Πακιστάν. Πρέπει οι θρησκευτικές μειονότητες να μπορούν και αυτές να συμμετέχουν στα κοινά και πρέπει να μπορούν να τελούνται όλες οι θρησκευτικές εορτές δεν υπάρχει κανένας νόμος ακόμη στο Πακιστάν που να μιλάει για την εγγύηση των ελευθεριών των μειονοτήτων. Υπάρχει η περίπτωση ετερόδοξο ζεύγος που ακούμπησε το Κοράνι να καταδικαστεί. Πρέπει λοιπόν φυσικά να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Πακιστάν και οι πολίτες του έχουν, πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα σε ό,τι μειονότητα και να ανήκουν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με ό,τι υπόθηκε προηγουμένως για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Πακιστάν. Ιδιαίτερα θα ήθελα να θέσω το θέμα των διώξεων των Αχμαντία Πρόκειται για διώξεις, για δολοφονίες καθαρά. Και αυτό συνεχίζεται και σήμερα παρά το γεγονός ότι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι τωρινοί υποσχέθηκαν βελτιώσεις που όμως δεν πραγματοποιήθηκαν. Οι διώξεις συνεχίζονται και νομίζω καιρό είναι πια η διεθνής κοινότητα μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξυπνήσει και να παρέμβει για να καταδικαστούν αυτές οι διώξεις και οι διωγμοί. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπέλντερ για την ομάδα του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν ιδρύθηκε το κράτος του Παγιστάν το 1947, ναι. ο, ε, ο ιδρυτής έλεγε ότι θα πρέπει όλοι οι πολίτες ε, να είναι ίσοι, έλεγε ο Τζίνα τότε, ανάλογα, ε, ανεξάρτητα από ε, την θρησκεία τους. Το Πακιστάν όμως έχει 15 εκατομμύρια χριστιανούς που τους καταπιέζουν αγρίως. Και μέχρι την πρωτεύουσα, το Ισλαμαμπάτ. Και επιπλέον το νομικό σύστημα ε, διατηρεί σε μειονεκτική θέση τους χριστιανούς. Έχουμε μια υφέρπουσα Ισλαμοποίηση, ένα εξισλαμισμό από τα τέλη του 70 της κοινωνίας. Και αυτό σημαίνει ότι είναι εις βάρος της χριστιανικής κοινότητας του Πακιστάν. Συγκεκριμένα έχουμε μαρτυρίες και το, νόμο για τη βλασφημία του 1980 και τα νομικά εργαλεία που θέτουν εκτός νόμου τους χριστιανούς. αν θέλει να ακούσει ως μάρτυρα ένα χριστιανό, ένας δικαστής, αυτό μετράει ε, ως μαρτυρία το μισό από ένα μουσουλμάνο. Και ε, το θέμα της βλασφημίας είναι πολύ σοβαρό και σχέση με το Κοράνι και με τον προφήτη και μπορεί να ε, επιβληθεί μέχρι και θανατική ποινή. Θα πρέπει ε, να ε, προστατεύονται οι χριστιανοί και οι μη μουσουλμάνοι από το να καταλήγουν σε ε, κελιά να περιμένουν πότε θα εκτελεστούν. Χρόνια ολόκληρα παραμένουν ε, στη φυλακή χωρίς καμία διαδικασία, χωρίς δίκη χριστιανοί παρακαλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, συνδέει οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας και βοήθειας με το ε, Πακιστάν ε, με την άρση αυτών των καταστάσεων εις βάρος των θρησκευτικών μειονοτήτων. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ερχόμαστε στις μεμονωμένες τοποθετήσεις. Η κυρία Αντρική είναι πρώτη για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το Σύνταγμα του Πακιστάν κάνει διάκριση μεταξύ μουσουλμάνων και μη μουσουλμάνων. αυτό συνιστά διάκριση με βάση τη θρησκεία. Είναι πολύ σημαντικό να θυμίσουμε εδώ ότι το Δεκέμβριο του 2009 ο ε, Αλή ε, ε, ο, Αζερτερή, ο πρόεδρος, είπε ότι οι μειονότητες έχουν το δικαίωμα να έχουν ίση μεταχείριση. Δυστυχώς όμως ανεξάρτητες μελέτε και έρευνες ε, έχουν αποδείξει ότι δεν ισχύει αυτό στην πράξη. Δεν υπάρχουν ούτε ε, αστικές ελευθερίες, ούτε ίσες ευκαιρίες, ούτε στην απασχόληση, ούτε στην πολιτική εκπροσώπηση. Και παντού ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειε τώρα, δεν έχουμε χρόνο, αλλά μα ανησυχούν πολύ αυτά που ακούμε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω επίση και μία αντίφαση μεταξύ της δέσμευσης κυβέρνησης του Πακιστάν ε, και ε, του ρόλου που παίζει στον ε, Οργανισμό Ισλαμικών Κρατών και στα Ηνωμένα Έθνη. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν θα ήθελα να θυμίσω τα συμπεράσματα του Νοεμβρίου της 16ης Νοεμβρίου του 2009 του Συμβουλίου για την προστασία των προσώπων, των ατόμων και των ομάδων ως προς τις διακρίσεις ε, κατά τις θρησκείες. Ευχαριστώ. Σας υπενθυμίζω ότι θα μας λείψει ο χρόνος σήμερα και όποιος ξεπερνάει αφαιρεί χρόνο από τους υπόλοιπους του ιδίως για την οφθαλμοθυρία. Ο κύριος Τσαρνέτσκι. Κοιτάξτε, Όπως λένε στην Αμερική δεν υπάρχει δωρεάν φαΐ. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε δωρεάν. Τα 200 εκατομμύρια ευρώ δεν μπορούν να μην έχουν κανένα αντίτιμο. Πρέπει να απαιτήσουμε το σεβασμό ορισμένων προτύπων και διεθνών αρχών που για μας είναι σημαντικές πολιτικές αρχές και που θα θέλαμε να σεβαστεί και το Πακιστάν όπου διώκονται άνθρωποι επειδή απλώς δεν έχουν την ίδια θρησκεία. Αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Γίνεται λόγος και στην Ευρώπη για μειονότητες ε, θρησκευτικές σημεί ε, και στην Ευρώπη φυσικά πρέπει να σεβόμαστε τις μειονότητες και στο Πακιστάν όμως τη χριστιανική και άλλες μειονότητες. Δεν είναι φυσικά το μόνο πρόβλημα της χώρας αυτής, όπου υπάρχει η πολιτική αστάθεια εδώ και πολλά χρόνια. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε δύο σημαντικά θέματα όσον αφορά την κατάσταση στο Πακιστάν. Το ένα είναι ότι είναι στρατηγικό εταίρο στην καταπολέμηση τη τρομοκρατία και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε την ε, ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Το άλλο γεγονό είναι ότι στο Πακιστάν υπάρχει επικρατή διαφορετική στάση απέναντι στι εθνοτικέ και θρησκευτικέ μειονότητε από αυτό που ισχύει στην Ευρώπη ή στις άλλες ανεπτυγμένες δημοκρατίες. Η Ευρώπη δεν μπορεί να εθελοτυφλεί αν ε, παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα χονδροειδώς. Γι' αυτό και θα πρέπει να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας ακόμα και αν πρόκειται για ένα στατηγικό εταίρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να θεωρηθεί αξιοπιστή όταν ε, ζητά λογαριασμό από τρίτε χώρε, όταν μπορεί να λύσει πρώτα τα δικά της προβλήματα για τις εθνοτικέ και θρησκευτικές μειονότητες ε, εντός Ένωσης. Ε, μία από τις ε, προτεραιότητε της Ένωση είναι να προστατεύει τις εθνοτικέ και θρησκευτικέ μειονότητες και θα πρέπει να τις εφαρμόζει η ίδια καταρχήν. Μόνο μετά μπορούμε να ζητήσουμε λογαριασμό από τους εταίρους μας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι το Πακιστάν ε, κατα... πολεμά μαζί με διεθνείς εταίρους είναι τρομοκρατία. Ωστόσο δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στα άλλα προβλήματα που ε, υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, όπως η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτών των θρησκευτικών και ε, μειονοτήτων. Τακτικά ακούμε μαρτύρια ακόμα και δολοφονίες χριστιανών. Τους καίνε ζωντανού μόνο και μόνο επειδή είναι χριστιανοί. Ακόμα και τα παιδιά καίνε. Μα γιατί συμβαίνει αυτό σε μια χώρα που ε, παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Συμβαίνει διότι οι αρχές του Πακιστάν έχουν συμβάλει στην ε, κατάσταση που ισχύει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Η νομοθεσία για τη βλασφημία παραδείγματος χάρη και το γεγονός ότι οι αστυνομικές δυνάμεις ε, δυσλειτουργούν είναι πράγμα το οποίο θα πρέπει σαφώς να κρατήσουμε σταθερή θέση. Κάστλερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Παγκοσμίω, 75 με 80% των διοκόμενων είναι χριστιανοί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο. Η ανεξιτρισκεία είναι βασικό στοιχείο τη πολιτική μα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό λυπούμε που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συχνά τα κάνουν πλακάκια αριστεροί και αριστεροφιλελεύθεροι και αποσιωπούν ε, τη μοίρα των χριστιανών. Χαίρομαι ε, που σήμερα αντιδρούμε γιατί η κατάσταση είναι φρικτή στο Πακιστάν και θα κάνουμε κοινό ψήφισμα από τα 156 ε, εκατομμύρια το κατοίκον, 95% είναι μουσουλμάνοι, 3% χριστιανοί και 2% Ινδουιστές. Ως χριστιανός θα ήθελα να μιλήσω για τους χριστιανούς του Πακιστάν που διώκονται σφοδρά. Όποιος επιτρέπει τη βία κατά των χριστιανών θα πρέπει να λάβει την απάντηση του πολιτισμένου κόσμου. Γι' αυτό θα πρέπει και στην οικονομική συνεργασία να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κριτήριο και τέτοιο στο μέλλον και ενδεχομένως να έχουμε και κυρώσεις. Ευχαριστώ. Παίρνουμε τώρα στη διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑ, αυθόρμητε τροποθετήσει. Έχω πολύ περισσότερα αιτήματα από εκείνα που μπορούμε να ικανοποιήσουμε. Επειδή έχουμε μόνο δύο λεπτά, θα πάρω τέσσερι τέσσερις ομιλητές. Πρώτος ο κύριος Γκάλε. Ναι, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι κάθε χώρα θα πρέπει να κρίνεται και με βάση την προέλευσή τη και την αφετηρία τη και ε, πώ εξελίσσεται η κατάσταση και αν πηγαίνει προς την ορθή κατεύθυνση. Εγώ ήμουν επικεφαλή των παρατηρητών τη Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από δύο χρόνια τις εκλογές και έκανα και κάποιε συστάσει. Και χαίρομαι που η χώρα αυτή ε, κατέβαλε προσπάθειε να εφαρμόσει τι συστάσει αυτέ, Για παράδειγμα την κύρωση του Διεθνού Συμφώνου για τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα. Ε, μεταξύ δεν την έχουν μόνο υπογράψει, την έχουν κυρώσει κιόλα ή τη σύμβαση κατά των είναι καλό τώρα πλέον που υπάρχει και υπουργό που ασχολείται ακριβώς με θέματα μειονοτήτων ε, ε, από το χαρτοφυλακείο, ε, χαρτοφυλάκιο του, είναι αρμοδιότητά του να καταπολεμά τις διακρίσεις. Αναφέρθηκε η μειονότητα των, των που έχουν ε, ε, χωριστούς εκλογικούς καταλόγους. Καλό θα ήταν να μπουν στους γενικούς καταλόγους για τις εκλογές, για να τερματιστεί αυτή η διάκριση. Ευχαριστώ. Uh, now, κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ότι συνήθισα και εγώ την εβδομάδα που μας πέρασε τον Υπουργό Μειονοτήτων του Πακιστάν. Και είμαι και εγώ πεπισμένη ότι προσπαθεί να βρει κάποια λύση και να συμφωνήσουν όλες οι μειονότητες. Αλλά ούτε εκείνο μπορούσε να απαντήσει, μπόρεσε καλύτερα ε, να απαντήσει στην ερώτησή μου γιατί το Πακιστάν στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών έχει αυτή τη στάση. Γιατί ε, συμφώνησε με τις άλλες Ισλαμικές χώρες ε, και ε, δεν μπορεί να προχωρήσει προς την κατέθεση της ανεξιθρησκείας και της προστασίας των θρησκευτικών ελευθεριών και την προσέγγιση των θρησκευτικών ομάδων. Νομίζω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε τέτοιου είδους νέοι κανόνες να επικρατήσουν και στα Ηνωμένα Έθνη πλέον και να τηρούνται. Η κατάσταση στο Πακιστάν αλλάζει διαρκώς και χρειάζεται να το παρατηρούμε πολύ προσεκτικά ώστε να μην ε, προβούμε σε σφάλματα. Είναι θετικό το ότι η κυβέρνηση έλαβε μέτρα για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των μειονοτήτων, όπως για παράδειγμα το 5% ποσόστοση για τις ε, θέσεις του δημόσιου τομέα. Επίσης ε, θα κρατήσουν ε, θέσεις για τους ηλικιωμένους και τις γυναίκες. Ωστόσο, θα πρέπει κάτι να γίνει για την νομοθεσία περί την λογοκρισία καθώς και τις διώξεις που ακόμα και τις δολοφονίες σε μελών ε, ομάδων μειονοτήτων. Ο ποινικό κώδικας επίσης θα πρέπει να αλλάξει, καθώς και η θανατική ποινή θα πρέπει να καταργηθεί. Δεν μπορούμε την 21ο αιώνα να επιτρέπουμε να θανατώνονται άνθρωποι για... επειδή βλασφήμισαν. Η κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι προηγούμενες εκλογές στο Πακιστάν σηματοδότησαν μια επιστροφή στη δημοκρατία. Δυστυχώς όμως, μερικές εβδομάδες μετά άρχισαν οι δολοφονίες. Η δολοφονία μάλιστα τη ηγέτιδος του Λαϊκού Κόμματος στο Πακιστάν. Η κυβέρνηση ζήτησε μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα που προτάθηκαν ήταν θετικά όπως διαπολιτισμικός διάλογος και η ποσόστοση 5% μειονοτικών για τις δημόσιες θέσεις καθώς και σεβασμός μη μουσουλμανικών εορτών. Επίσης δέχτηκε η κυβέρνηση να δοθούν και θέσεις βουλευτών σε μειονοτικούς. Και επίσης ο ρόλος του Πακιστάν είναι σημαντικός στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη για προς όσους δεν μπορώ να δώσω το λόγο. Τώρα όμως θα μιλήσει ο Επίτροπος σύντομα. Κυρίες και κύριοι βουλευτέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση των μειονοτήτων στο Πακιστάν και του οποίου το Σύνταγμα αναγνωρίζει την ανεξιθρησκεία και προβλέπει ότι το κράτος προστατεύει τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Το Πακιστάν έχει σημειώσει προόδους τελευταία με τροποποιήσεις του συντάγματος. Άλλαξε το ρόλο και τη σημασία του Κοινοβουλίου. Ζητήθηκε μεγαλύτερο σεβασμό στα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημιουργήθηκε Υπουργείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υπουργείο Μειονοτήτων και αυτή τη στιγμή δημιουργεί ένα ανεξάρτητο Συμβούλιο Μειονοτήτων. Εξάλλου συνυπέγραψε και το σύμφωνο για τις πολιτικές ελευθερίες και την καταδίκη των βασανιστήριων και άλλων απανθρώπων μεταχειρήσεων. Όλα αυτά είναι θετικά εφόσον βέβαια εφαρμοστούν πράγματι. Πρέπει το Πακιστάν βέβαια να συνεχίσει τις προσπάθειές του, να πολλαπλασιάσει τις προσπάθειές του σεβασμού των, των θρησκευτικών τίτων μεταξύ των οποίων και των χριστιανών. Η διεθνή φήμη του Πακιστάν έχει αμαυρωθεί από γεγονότα όπως εκείνα τα περσινά στην Κόγια όπου εκάησαν ζωντανοί χριστιανοί από εξτρεμιστάς μέσα σε μια εκκλησία μάλιστα Επίσης σημειώθηκαν επιθέσεις κατά Σιητών, μεταξύ Σιητών και Αχμαδιστών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συστηματικά χρησιμοποιεί ως μέσω συνεννόησης τον πολιτικό διάλογο. Θέτει τα προβλήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επίσης κάνει και διπλωματικές χειρονομίες. Από το 7 άρχισε διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα πλαίσια της ε, διαλόγου συμφωνίας μεταξύ του Πακιστάν που συνεχώς αναφέρεται και σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο διάλογο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε επιμένει τα δικαιώματα των μειονοτήτων να γίνονται σεβαστά. Στα πλαίσια επίσης του διαλόγου αυτού για τα ανθρωπίνα δικαιώματα η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης τακτικά τονίζει προς την κυβέρνηση του Πακιστάν ότι πρέπει να αλλάξει η εφαρμογή του νομοσχεδίου για τη βλασφημία Ξέρω ότι έχουν καταδικαστεί και μουσουλμάνοι για αυτόν τον λόγο, αλλά παρόλα αυτά συνήθως το νομοσχέδιο αυτό εφαρμόζεται κατά μειονοτικών και ότι έχουν υπάρξει και ψεύτικες κατηγορίες. Η τελευταία συνεδρία της Μικτής Επιτροπής έγινε στις 25 Μαρτίου του Ευαγγελισμού και συζητήθηκαν εκεί πάλι θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλής διακυβέρνησης καθώς και το θέμα των μειονοτήτων. Εμείς δεν διστάσαμε να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει τα, όλα αυτά τα θέματα να τα ξαναθήξει και στην επόμενη διάσκεψη με το Πακιστάν στις 4 Ιουνίου. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού του Πακιστάν δεν έχει πρόσβαση στην παιδεία μέσω των βοήθειας που χορηγούμε εμείς δίνουμε προτεραιότητα στην πρόσβαση στην παιδεία για όλους. Ελπίζω ότι μέσω πρόθεσμα θα οδηγήσουν όλα αυτά σε μεγαλύτερη ανοχή και ανεξιθρησιουκία. Σας κατευχαριστώ όλους και όλες. Και εμείς σας κατευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Εφτά ψηφίσματα έχουν κατατεθεί. Έληξε εδώ η συζήτηση και η ψηφοφορία τους θα γίνει στο τέλος της συζήτησης. Επόμενο θέμα είναι η κατάσταση.